Hanno votato tutti? Ψήφισαν όλοι. Έχουν ψηφίσει και οι ψηφολέκτε. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας, ε, οι ψηφολέκτες θα πάνε στην αίθουσα R11 για την ε, ε, καταμέτρηση. Αναστέλλεται η ε, συνεδρίαση θα χτυπήσει το κουδούνι και θα ανακοινωθεί στις οθόνες ε, ε, πότε θα ξαναξεκινήσουμε.